Good morning, dear colleagues. Can you please sit down so that we start? Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. So, good morning, everybody. Let me start. Uh, Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Επιτροπή των Οικονομικών Τη οικονομική και Νομισματικής πολιτική. Έχω συνοηθεί με τον πρόεδρο και θα κάνει εκείνο τι ανακοινώσει όταν έρθει. Περνούμε λοιπόν κατευθείαν στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Ελέγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Σας καλωσορίζω. Έχουμε και κάποια επέτειο σήμερα του κοινού ελέγχου κατεξουδότηση πράξεων και εκτελεστικών μέτρων. Έχουμε λοιπόν εορταστική εκδήλωση με τον ε, έλεγχο αυτών. Ξέρετε ότι μερικές φορές ε, λαμβάνονται αποφάσεις ε, για πολύ περίπλοκες πράξεις και πιστεύουμε ότι αυτός ο έλεγχος των κατεξουδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων είναι πολύ σημαντικό και αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Με χαρά βλέπω την αθρώα προσέλευση αυτό το σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. 1η Ιανουαρίου του 2018 λοιπόν ε, τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός 11 για, τα, ε, για τους δείκτες αναφοράς σε σχέση με, τις, ε, με τα χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά μέσα. Περνάει μια συμβουλευτική φάση η ΕΣΜΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να μετατρέψει σε εκτελεστικές πράξεις τα κείμενα με βάση και τις προτάσεις μας. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε τα πιο σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με, αυτούς, ε, με αυτή την πράξη, τον ορισμό δηλαδή της διάθεσης στο κοινό, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια των ε, δικτών αναφοράς, μεταφατικές διατάξεις, εισαγόμενα δεδομένα και ορισμούς σχετικούς με τους διαχειριστές. Έχουν διατεθεί τα σχετικά έγγραφα και καλωσορίζω τον Φάσιο Πλάτα από την ΕΣΜΑ και τον κύριο Ρούντερ από την ΦΙΣΜΑ, Γενική Διεύθυνση. Θα μας κάνουν τις παρουσιάσεις. Σε πέντε λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Και μετά θα ακούσουμε εισηγητές και οδησηγητές και διαδικασία κατσιδιάης στη συνέχεια. Κύριε Πλάντα, εσείς, από την ΕΣΜΑ παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μας προσφέρετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα μέτρα επίπεδου 2 που έχει προβλέψει η ΕΣΜΑ. Πριν σας δώσω και τις ε, θέσεις της ΕΣΜΑ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή και σκιώδη συγητέ ισχυώδεις ηγητέ για το ενδιαφέρον στη συνεχιζόμενη αυτή διαδικασία και την επικοδομητική στάση. Είναι ευπρόσδεκτη αυτή η γραμμή επικοινωνία και η συνεργασία με, τη με την ομάδα των διαπραγματεύσεων και το προσωπικό. Δύο τύποι λοιπόν μέτρων τύπου 2. 10 Νοεμβρίου 2016 τεχνικές προτάσεις, τεχνικές συστάσεις, διάφοροι τομείς, διευκρινήσεις ορισμιών, των οποίων ορισμένους αναφέρατε κι εσείς μέτρηση της αξίας αναφοράς, του δίκτυα αναφοράς, ε, ιδιαίτερη σημασία δίκτες αναφοράς και ε, δίκτες αναφοράς τρίτων κρατών, μεταβατικές διατάξεις. Επίσης, ε, τεχνικές προτάσεις το Μάρτιο του 2017 με την εποπτεία πάλι θευσιμότητα των ε, δεδομένων εισόδου, διαφάνεια, κώδικα συμπεριφοράς, διαχείριση, διακυβέρνηση, εποπτεία των συνεισφερόντων, ποιοτικά κριτήρια για, σημαντικά, για σημαντικούς δείκτες, format για, τους, για τα σημαντικά και μη σημαντικά ε, σημαντικούς και μη σημαντικούς δείκτες, περιεχόμενο, ε, συστήματα πιστοποίησης αναγνώρισης, περιεχόμενο, εφαρμογή ελάχιστο περιεχόμενο συνεργασίας και διευθετήσεων μεταξύ ΕΣΜΑ και αρμόδιων αρχών. Τεχνικές προδιαγραφές επίσης από την Δευτέρα Ιουνίου με τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις έχουν διατυπωθεί για τις αρχές εποπτείας έτσι ώστε και για τις εκτελεστικές αρχές έτσι ώστε οι δείκτες να λειτουργούν σωστά με πλήρη επεξεργασία του τρόπου διατύπωσης των δικτών, επαλήθευση των νέων εποπτικών δραστηριοτήτων του διαχειριστή, ε, ελαχιστοποίηση του, της πιθανότητας παραποίησης, διαχείριση σωστή ισότιμο πεδίο σε όλα τα κράτη-μέλη για την πιστοποίηση και αδειοδότηση των δικτών. Η ΕΣΜΑ συνιστά τα δεδομένα που συλλέγονται από τρέχουσες και μελλοντικές ε, δομές αναφοράς όπως ΜΙΑΡ και ΜΙΦΙΤ και λοιπές να αξιοποιούνται στην κατάρτιση των δικτών όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διαβούλευση και το ενδιαφέρον που εξεδήλωσαν οι ε, διάφοροι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς. Με βάση το πρώτο, τους στόχους των μέτρων ε, τύπου 1 και 1 και επίπεδου 2, μιλούμε για την ακαιρεότητα και την επαληθευσιμότητα των δικτών. Μέτρα αναλογικά επίσης έχουν εισαχθεί σε σχέση με τους ιδιαίτερα σημαντικούς δείκτες τεχνικά χαρακτηριστικά με μια ολιστική προσέγγιση που θα περιορίσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τον διαχειριστή των δικτών και επίσης καθήκοντα που έχει αναλάβει η ΕΣΜ, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω, όπως προκύπτουν από τον κανονισμό και να σας πω και τι έχουμε κάνει. Διατηρεί λοιπόν μητρό των αδειοδοτηθέντων διαχειριστών η ΕΣΜΑ, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς μόνο εάν ο διαχειριστής ή ο ίδιος ο δείκτης περιλαμβάνονται στο μητρό μπορούν να χρησιμοποιούνται. Έχουμε επίσης πόρους, ε, έχουμε περιορισμούς ως προς τους πόρους της πληροφορικής και μηχανογράφησης ε, και έχουμε αντιμετωπίσει αυτούς τους ε, περιορισμούς ικανοποιητικά έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι από 1η Ιανουαρίου του 2018 να, τους, να θέσουμε τα συστήματα σε λειτουργία. Σημαντική εποπτική σύγκληση επίσης εξασφαλίζεται με εναρμονισμένους κανόνες, με τη σύγκληση των εποπτικών δράσεων και όπως άλλωστε αναφέρεται και στο μεθοδολογικό πλαίσιο για την υποχρεωτική συνεισφορά στους κρίσιμες σημασίες ε, δείκτες αναφοράς ε, έχουμε ορίσει και τις ειδικέ εξουσίες των επιτροπών, σημαντικό επίσης ε, εργαλείο για την εξασφάλιση της συνέπειας και της σύγκλησης, που δεν είναι πάντως απαραίτητα ένα μέτρο το οποίο σκοπεύουμε να ενεργοποιήσουμε. Ελπίζουμε ότι θα χρειαστεί σπάνια να αξιοποιηθεί και ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Λάουντρουπ από την Αυμόδια Γενική Διεύθυνση μέχρι 5 λεπτά. Αν θέλετε να μιλήσετε περισσότερο, Είστε ελεύθερος. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι παρόν και να σας παρουσιάσω τις αρχικές μας προτάσεις. Συγχαρητήρια καταρχάς για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε η ΕΣΜΑ. Δύο ομάδες δουλειάς έχουν ολοκληρωθεί. Καταρχάς η κατεξουσιοδότηση πράξης και μετά τα λεγόμενα RTS. Καταρχάς, έχουμε ολοκληρώσει εμείς την αξιολόγηση των κατεξιοδότηση πράξεων, έχουμε ενημερώσει και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε συλλέξει τα σχόλια από τους νομικούς μας συμβούλους και τώρα θα περάσουμε άμεσα στο επόμενο στάδιο, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μια δημόσια διαβούλευση μηνιαίας διάρκειας όπως προβλέπεται από τον κανονισμό για την κατεξουσιοδότηση πράξη. Βλέπετε λοιπόν ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία σύμφωνα με την αρχή της διαβούλευσης. Δεν θα υπάρξουν πολλές αλλαγές, νομίζω δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, ίσως να υπάρξει μια τεχνική αναδιατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων εμείς δεν είχαμε την πρόθεση με τα περισσότερα από όλα αυτά να αποκλίνουμε από αυτά τα οποία λέγει η ΕΣΜΑ. Τώρα αν οι δικηγόροι μας, οι νομικοί μας σύμβουλοι αλλάξουν κάποιες από τις ε, διατυπώσεις θα σεβαστούμε γενικά τις βασικές γραμμές τις οποίες προτείνει η ΕΣΜΑ. Θα περάσουμε ίσως σε λίγο περισσότερη λεπτομέρεια στα λεγόμενα κομβικά για μας θέματα το θέμα της διαθεσιμότητας σαν παράδειγμα όταν υπάρχει ένας τέτοιος δείκτης ε, να είναι διαθέσιμος στο κοινό. Αν υπάρχουν τώρα για τέτοιου είδους διατυπώσεις κάποιες ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας. Μία δεύτερη σημαντική έννοια η οποία περιλαμβάνεται στην κατεξουσιοδότηση πράξη είναι οι αντικειμενικές αιτίες για παροχή τέτοιου είδους δικτών σε αρχές και υπηρεσίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπει μια διαδικασία η οποία ελέγχει το αν είναι αντικειμενική η λόγοι για την δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου τεχνικού δίκτυ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι ιστορικά μέχρι τώρα στο παρελθόν οι δείκτες κυκλοφορούσαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή είναι η βασική, αν θέλετε, γραμμή και η παράδοση την οποία έχουμε ε, για όλες τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε κάποιες περαιτέρω ερωτήσεις. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι σε επίπεδο χρονισμού εμείς ε, έχουμε με αυτή την πράξη ε, νομίζω την δυνατότητα για ένα σταθερό, ασφαλές, αναθεωρημένο νομικό δεσμευτικό κείμενο. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο Φαμπρίτσιο. Είναι σαφές ότι είναι ε, μεγάλο σε μέγεθος, αυτό θα πρέπει ίσως να το επανεξετάσουμε, το έχω παραδεχθεί και στο παρελθόν αυτό θα περάσει από μια νομική μεταρρύθμιση. Θα υπάρξει μια επί της μεταρρύθμιση σε επίπεδο νομικό και θα ακολουθήσει μια γλωσσική αντίστοιχη. Πάντως είπαμε ξεκινάει το κείμενο αυτό από την επόμενη εβδομάδα να είναι διαθέσιμο σε επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης. Λίγο μετά τον Ιούνιο θα κλείσει η διαδικασία διαβούλευσης Ελπίζω, ε, νομίζω ότι θα υιοθετηθεί επίσημα μετά ε, τα καλοκαίρι γιατί είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο τον μήνα Αύγουστο. Μετά θα περάσει έτσι και αλλιώς από τη διαδικασία περίοδου ελέγχου και αυτό είναι παραδεκτό και θα υπάρξει πάλι ένας μήνας διαβούλευσης. Πάντως είναι σαφές ότι και οι έννοιες είναι ξεκάθαρες τώρα πλέον και η διαδικασία είναι γνωστή και ανοιχτή και είμαι βέβαιος ότι το περιεχόμενο και η ουσία είναι εδώ μαζί μας τώρα και θα εξεταστεί από την επόμενη εβδομάδα. Έχει έτσι και λιώς την περίοδο ελέγχου την κοινοβουλευτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να την χρησιμοποιήσει εφόσον το επιθυμεί έτσι ώστε να προλάβουμε τις διαδικασίες που θα μας δώσουν την εφαρμογή του κανονισμού αυτού από τον Ιανουάριο του 2018. Δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια να συμπέσουν χρονικά τα αποτελέσματα της εξέτασης από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ημερομηνία θέση σε ισχύ ε, ε, ε, θέση σε ισχύ της συγκεκριμένης πρόταση, γιατί έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή είναι γνωστά. Η κόρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω και την ΕΣΜΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη την δουλειά που έχει γίνει και βλέπω ότι έχετε εργαστεί πολύ σκληρά αλλά ελπίζω να μην υπάρξει πρόβλημα επικάλυψης το, της περίοδου ελέγχου και της αρχής της ε, εφαρμογής. Λοιπόν, όταν θέλουμε να ελέγξουμε πρέπει να ξέρουμε ποιος ήταν ο στόχος αυτής της νομοθεσίας. Γιατί βλέπουμε σε λεπτομέρειες, αλλά η βασική αρχή θέλουμε να μην υπάρχει ενδεχόμενο επηρεασμού. Γι' αυτό εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να υπάρχει σωστή εποπτεία, περισσότερη διαφάνεια, αλλά είπαμε επίσης ότι πρέπει να είναι και αναλογική. Γι' αυτό είχαμε τις δύο κατηγορίες της κρίσιμης και μη κρίσιμης κατάστασης. Τώρα είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση, αλλά η αρχή της αναλογικότητας βεβαίως εξακολουθεί να ισχύει. Βεβαίως πρέπει να είναι και λειτουργικό το σύστημα. Δεν θέλουμε να είναι υπερβολικά αναλυτικό. Όσο λιγότερη γραφειοκρατία γίνεται. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Και έτσι θα εξετάσουμε όλες τις κατεξοδότηση πράξη και τα RTS Επίσης, δεν θέλουμε να υπάρχει επικάλυψη με άλλους κανονισμούς. Θέλουμε δηλαδή να αποφύγουμε επικάλυψη, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, θέλουμε να αποφύγουμε αντιφάσεις ή συγχύσεις στους ορισμούς ή αλλού. Τώρα, τι προτάσεις περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να είναι λειτουργικό αυτό το οποίο εγκρίνουμε. Δεν θέλουμε να, προ... προκύψει στρέβλωση των αγορών. Άρα χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος. Είναι πολύ σημαντικό. Εφόσον έχουμε ήδη καθορίσει την ημερομηνία και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα φροντίσετε ότι θα αποφευθεί κάθε ούτως ώστε να αποφευθεί κάθε στρέβλωση των αγορών. Δημιουργούμε βέβαια νέες τιμές αναφοράς, ε, ακόμη και καθημερινά, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να μπορέσει να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία των αγορών. Πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό. Βεβαίως είναι και θέμα ερμηνείας των κανόνων, αλλά η δική μας λοιπόν ερμηνεία, να καταστήσω σαφές, είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρξει στρέβλος των αγορών. Τώρα, πεδίο εφαρμογή. Θα θίξω ορισμένα θέματα όχι κατά ανάγκη από τα πιο σημαντικά στα λιγότερο, αλλά γενικά. Τώρα, για το πεδίο εφαρμογή. Έχουμε την εντύπωση ότι έχει επιτύχει τη σωστή ισορροπία η ΕΣΜΑ με τις προτάσεις της. Αλλά πάντα βεβαίως, ε, τα πάντα είναι βελτιώσιμα. Δηλαδή, για το κείμενο τεχνικών συμβουλών για την έκδοση και χρήση, τότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ούτως ώστε τα περιθώρια ε, να είναι σαφή. στο επίπεδο 1 λέμε ότι τα περιθώρια, το clearing και τα λοιπά δεν θα βασιστούν σε τιμές αναφοράς ή σε δείκτες αναφοράς. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι οι εξαιρέσεις για τις δημόσιες αρχές, ε, τις ε, ενωσιακές και μη ενωσιακές τράπεζες, ε, τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συμβάλλουμε στον καθορισμό των δικτών τους. Και αυτό συνάδει με τις ιδεολογικές μας σκέψεις 14, 15, 16 και 19. Είναι ζωτική σημασία. Γιατί η, τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών χρησιμοποιούνται πολύ. Άρα οι δικοί τους ε, οι δείκτες αναφοράς πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι δικοί μας. Τώρα υπάρχει και ένας άλλος κανονισμός, όπως ξέρετε, που ήδη λειτουργεί. Αφορεί, ε, αφορά τις διαδικασίες over the counter που γίνονται μέσω ε, των εσωτερικών συστημάτων. Θέλουμε λοιπόν να ε, συμβαθεί η λειτουργία τους με την οδηγία MIFID 2. Τώρα, για τις τρίτες χώρες. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Από την πλευρά των ενωσιακών χρηστών των δικτών αναφοράς, πρέπει να καθοριστεί σαφές ότι η αναγνώριση ενός μη ενωσιακού διοικητή του επιτρέπει να εφαρμόσει τις αρχές ΙΟΣΚΟ ε, ΑΙΟΣΚΟ και άρα να υπάρξει συμμόρφωση. Βασιζόμαστε πάντως αυτό και οι προϋποθέσεις BMR εφαρμόζουν ε, τα κριτήρια IOSCO. Αυτό θα πρέπει να το ελέγχουν οι εθνικές αρχές με βάση τα αποτελέσματα και όχι σύγκριση γραμμή προς γραμμή. Δεν είναι αυτό το πνεύμα της νομοθεσίας που θέλαμε να ισχύσει. Τώρα ίσως είναι δευτερεύον, αλλά έχει τη σημασία του. Τα ρυθμιστικά τεχνη, οι ρυθμιστικές τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι υποχρεωμένες να δώσουν πληροφορίες σε επίπεδο α στο οποίο δεν λειτουργούν, στο οποίο δεν εφαρμόζονται. Είναι προφανές ίσως, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να μην υπάρχει μία αντιμετώπιση για όλες τις καταστάσεις. Για παράδειγμα, στον τίτλο 2 υπάρχουν ε, προϋποθέσεις, προδιαγραφές για τον κώδικα διοντολογίας. Ορισμένα εμφανίζονται στο ε, σχέδιο του κώδικα RTS. Πρέπει να υπάρχει σωστή διάκριση. Εάν υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα για διαφορετικά ε, διαδίκτες αναφοράς για μερικά βασικά εμπορεύματα. Ε, αλλά ίσως να έχουν και άλλοι συνάδελφοι σχόλιο, οπότε να σταματήσω εδώ. Εκ μέρου ε, του ΕΛΚ και ευχαριστώ κόρα, θα είμαι και ο πρέπει να μιλήσω εγώ. Είπε πολλά θέματα σοβαρά, σημαντικά και τεχνικά. Είμαι εγώ πιο γενικό. Πρώτα απ' όλα, είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή του Κοινοβουλίου Σκιώδη. Είχαμε πολλέ χρήσιμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνεχίζονται και ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα στο οποίο δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο είναι η επιλογή του χρονικού σημείου για τη δημοσίευση των προτάσεων μετά τις θερινές διακοπές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το μόνο που, πρέπει, που μπορεί να είναι βέβαιη η αγορά είναι ότι θα χρειαστεί να περιμένει. Και λυπούμε γι' αυτό, γιατί ήταν σαφές μέχρι πριν από λίγο το χρονοδιάγραμμα που θα, θα ακολουθούσαμε. Χάσατε χρόνο όμως ο λίγων εβδομάδων και αυτό οδήγησε σε αβεβαιότητα. Και το, πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα είναι να καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνουμε για να μπορεί να προσαρμοστεί. Εάν, το φτάσουμε σε αυτό το σημείο της αφήνειας των καθαρών κανόνων, δεν θα να κάνει κανονισμός και βέβαια του χρόνου για προσαρμογή. Γι' αυτό λυπούμε ιδιαίτερω για την καθυστέρηση αυτή. Και επί της ουσίας, τώρα, ανέφερε και η συνέλφωση νωρίτερα, δεν ήταν στόχος μας να επιβάλλουμε ένα κανονισμό ε, βαρύ και δυσκίνητο, αλλά έναν κανονισμό καλό που θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα με ορατότητα. Που θα εξασφάλιζε ότι ο πελάτης αλλά και ο χρήστης θα μπορούσε ανάλογα με την ανάγκη του να επιλέγει τους δείκτες αναφοράς το στηρίζεται. Αναλογικότητα ήταν η κύρια για μας ε, ιδέα και αρχή και χαίρομαι που η ΕΣΜΑ και η Επιτροπή έχουν αποφασίσει να ε, διατυπώσουν τις σχετικές προτάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την μεταφορά στην ε, χρήση, την διάθεση, τις διάφορες κατηγορίες δίκτων αναφοράς. Είπε και η ότι δεν θέλαμε πιο περίπλοκες κατηγορίες, αλλά το δεχόμαστε κατόπιν του τριμερούς διαλόγου και χαίρομαι που κάνετε και εσείς μια προσπάθεια για περιορισμό λίγο πολύ αφού υπάρχουν επικαλύψεις λίγο πολύ στα νομοθετήματα. Το μόνο που από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν είναι σαφές είναι αυτό που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις και ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ξέρω πως η ΕΣΜΑ έχει ζητήσει από την Επιτροπή να, καταστήσει, να καταστήσει σαφές πως ε, τόσο για τους ε, ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρόχους των υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφείς οι προθεσμίες και η μεταβατική περίοδος. Ο κύριος Μου Φερνάντες τώρα εκ μέρους και Δημοκρατών, πάλι ο Σκιώδης. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες για τις διαδικασίες εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού. Θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις. Στις 30 Μαρτίου η ΕΣΜΑ δημοσίευσε την πρόταση για τα RTS που περιλαμβάνουν ακριβώς, που είναι συνέπεια μάλλον της νομοθετικής αυτής ρύθμισης που έγινε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με μια ολόκληρη σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτούν περαιτέρω διευκρινήσεις. Θέλει τρει μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποδεχθεί ή όχι την ερμηνεία που δίδει η ΕΣΜΑ για τα RTS αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία στο τέλος Ιουνίου το πώς βλέπει την ερμηνεία την οποία δίδει η ΕΣΜΑ. Δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στην αποδοχή δικτών ή μάλλον τις διευκρινήσεις των δικτών και τον χαρακτηρισμό τους ως δικτών κρίσιμου επίπεδου. Στο εσωτερικό αυτής της ε, κατηγοριοποίησης λοιπόν ε, αυτών των κρίσιμων δικτών, των δικτών συγγνώμη, κρίσιμης σημασίας θα πρέπει να μας πει η ΕΣΜΑ τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις οι οποίες είχαν γίνει δεκτές και έχουν συμπεριληφθεί στον κανονισμό που έχει και αυτός γίνει δεκτό και είναι θα έλεγα υποχρεωτική η εφαρμογή τους σχετικά με το Euribor. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα παίξει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έτσι και αλλιώ ε, οι συμμετέχοντες θα είναι, υποχρεωτικοί να, είναι υποχρεωτικό να καταβάλουν την συγκεκριμένη αυτή να δεχθούν αυτήν την διαδικασία και αυτό δημιουργεί θέμα σε σχέση με την ανάπτυξη του Euribor Plus και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή του λόγω ακριβώς αυτής της υποχρέωσης συνεισφοράς, κάτι το οποίο για μια ακόμη φορά θα θέσει σε δύσκολη κατάσταση, σε πολύ δύσκολη κατάσταση τα πιστοτικά ιδρύματα τους επόμενους μήνες. Πώς λοιπόν αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράλυση, θα λέγαμε, του Euribor Plus ακριβώς μέσω της εφαρμογής ενός νέου δίκτυ κρίσιμης σημασίας. Τώρα για τις επιπτώσεις του Brexit, η τρίτη ερώτηση. Σε αυτό ε, έχουμε προβλέψει εδώ διαφορετικές επιλογές οι οποίες θα μας επιτρέψουν στο εσωτερικό της Ένωσης δικτών οι οποίοι να έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι επιλογές έχει ο κανονισμός. Ε, αναγνώριση δικτών, αποδοχή δικτών, απλή εφαρμογή ε, οι διαδικασίες αυτές είναι επαρκείς έτσι ώστε να μας επιτρέψουν στο μέλλον να χρησιμοποιούμε τους δείκτες του Ηνωμένου Βασιλείου, σαν παράδειγμα. Ή μήπως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο αναγνώρισης και πιστοποίησης. σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Μπορεί κάποιος ε, να μιλήσει εξ ονόματος των συντηρητικών. Τώρα βλέπω τον εκπρόσωπο των Πρασίνων, ο κ. Κίγκολτ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω το γεγονός ότι στην Επιτροπή μας όλο και περισσότεροι ντύνονται με πολύ χαλαρό τρόπο. Ακόμη και οι προσκεκλημένοι μας δεν φοράνε πια γραβάτα. Νομίζω ότι η ΕΣΜΑ όμως ακόμη είναι υπερβολικά καλοντημένη βλέπω ότι όντως ε, περνάμε σε πράσινο ντύσιμο. Ένα θέμα έχω όσον αφορά το καθεστώς τρίτων χωρών. Το έχουμε συζητήσει πολύ. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τις τρίτες χώρες εν ώψη των επικειμένων εξελίξεων. Και αυτή η συζήτηση επέδρασε και στην διατύπωση των μέτρων επίπεδου 2. Και δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε ποιοι δείκτες θα περιληφθούν ή δεν θα περιληφθούν για το καθεστώς των τρίτων χωρών. Και τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν και η ΕΣΜΑ για να αποδεχθούν τις ισοδύναμες εποπτικές αρχές. Και τι θα σημάνει αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο, το έχετε σκεφτεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις πολιτιστικές και για τις οικονομικές παρατηρήσεις σας. Τώρα, αν κάποιος άλλος συνάδελφος ε, θέλει το λόγο, υπάρχει χρόνος. Αν όχι, τότε θα τελειώσουμε και πιο σύντομα από ό,τι προβλέπαμε. Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της ΕΣΜΑ πρώτα απ' όλα για το μεταβατικό καθεστώς που ανέφεραν διάφοροι ευρωβουλευτές βεβαίως και θέλουμε να διευκρινίσουμε μέσω ερωταποκρίσεων την εφαρμογή των θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταβατική περίοδο αλλά θέλουμε να δούμε εάν η ερμηνεία μας ε, που συμφωνεί με αυτά που είπατε είναι αυτή την οποία είχε κατά νου ο νομοθέτης. Υπάρχει κάποια αναφορά σε δείκτες αναφοράς στη μεταβατική περίοδο. Εμείς θεωρούμε ότι οι μεταβατικές διατάξεις αφορούν τις διοικητικές αρχές και η αναφορά ε, στις, στους υπάρχοντες ε, δείκτες αναφοράς θα σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Εάν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία που κάνουμε, αυτό θα μας επέτρεπε οι υπεύθυνοι θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους να διατυπώνουν νέους δείκτες αναφοράς και δεν θα υπάρξει η διαταραχή που θα προέκυπτε από μια πιο αυστηρή ερμηνεία. Δηλαδή να βασιζόμαστε στις υπάρχουσες τιμές αναφοράς και όχι στην δραστηριότητα του διαχειριστή. Εάν οι συνομοθέτες συμφωνούν, τότε μπορούμε να διατυπώσουμε αυτή τη διευκρίνηση αλλά πείτε μας εάν συμφωνείτε ότι αυτή ήταν η πρόθεση του νομοθέτη. Γιατί έτσι τουλάχιστον εμείς ερμηνεύουμε την πρόθεση του νομοθέτη. Πολλές ερωτήσεις ε, απευθύνονταν περισσότερο στην Επιτροπή κανόνες για, για τις τρίτες χώρες αφορούν περισσότερο το κατά πόσο είναι κατάλληλο το υπάρχουν καθεστώς λόγω του Brexit. Οπότε είναι θέμα περισσότερο των συνομοθετών να δουν αν χρειάζεται αναθεώρηση. Δεν είναι θέμα δικό μας εφαρμογής δηλαδή. Δεν είναι θέμα τεχνικών προδιαγραφών. Για άλλα θέματα έχουμε εκφράσει την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικό καθεστώς για τις τρίτες χώρες. Και στα πλαίσια της ανθεώρησης του ESA ίσως να υπάρξουν εξελίξεις για τα θέματα αυτά. Αλλά όπως είπα είναι κυρίως θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τους συνομοθέτες. θα εργαστούμε βάσει το υπάρχον καθεστώ. Όσο για το θέμα του Euribor που αναφέρθηκε. Βεβαίως είναι θέμα. Ήδη ανακοινώθηκε ότι δεν λειτουργήσε όπως αναμενόταν το πείραμα Euribor Sin παρατηρούμε στενά ποιες άλλες εναλλακτικές θα μπορούσαν να υπάρξουν μαζί με την Κομισιόν και άλλες ρυθμιστικές αρχές όπως το SMA όπως ανακοινώσαμε στόχος μας είναι η μεταβατική περίοδος να είναι όσο δυνατόν λιγότερο επιβλαβής για την αγορά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πιο συγκεκριμένο γιατί πρέπει να αναλύσουμε ποιες άλλες εναλλακτικέ διαθέτουμε και τι επίπτωση θα είχαν. Αλλά παρατηρούμε στενά τη διαδικασία για να υπάρξει όσο το δυνατόν λιγότερη διαταραχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, όντως προς τις ερωτήσεις είχαν ε, στόχο την Επιτροπή. Πάντως ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, τα σχετικά με τη μετάβαση. Εύστοχα μου φαίνονται και λογικά, αλλά σε ακούσουμε την Επιτροπή και με το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα που θα φτάσει πιστεύω, μπορούμε να ξανακούσουμε την κόρα και άλλου σκιώδει, εάν σκοπεύουν να δευτερολογήσουν. Α ακούσουμε την Επιτροπή λοιπόν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον Σβέν Γκίγκολτ που αναγνώρισε ότι ερχόμαστε σε μια ε, πιο cool στάση. Είναι πιο δύσκολο να περάσει κανείς ε, τους ε, πολύ αυστηρούς είναι πιο εύκολο να περάσει κανείς τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας ε, στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λιγότερα πράγματα χρειάζεται να, να βγάλει κανείς, σακάκια κτλ. Και άρα μας διευκολύνει αυτό. Δεν θα έρθω βέβαια με τη ρόμπα, σας διαβεβαιώ, και τις παντόφλες. Τα παπούτσια απαιτούνται για να μπούμε μέσα. Μεταβατικά λοιπόν, μεταβατικά μέτρα. Το... Η ΕΣΜΑ ήδη ανέφερε ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση, μια προσέγγιση λογική και θα ήθελα και εγώ επί τη ευκαιρία να επιβεβαιώσω ότι στο άρθρο 51 προβλέπουμε την μεταβατική περίοδο σε δύο στάδια μάλιστα αναφέρεται στο 51.1 για τον πάροχο. Ο πάροχος βρίσκεται στην αγορά, έχουμε ένα δίκτυο αναφοράς και μπορεί, χρειάζεται μόνο να ζητήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2020 την άδεια. Αυτό έχει να κάνει με τη μεταβατική περίοδο που σχετίζεται με τον ε, πάροχο. δάλος ε, θα πρέπει να είναι λοιπόν μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, αυτό λέμε. Και στη δεύτερη περίπτωση, 51-2, εάν έχουμε την προσέγγιση με βάση το χρήστη, τη στιγμή της ε, υποβολής της αίτησης, όπως εξήγησε και ο Φαμπρίσιο, 1η Ιανουαρίου του 2018 με τη θέση της εισαγωγή του κανονισμού. Εάν υπάρχει ήδη ένας δίκτυς αναφοράς, μπορούν να το χρησιμοποιούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 οι αρχές. Επομένως έχουμε τον ίδιο τον ε, πάροχο ο οποίος θέλει να βγει στην αγορά με ένα προϊόν και μπορεί να αναβάλει την ε, αδειοδότηση μέχρι το 2020. Ιδάλλως όταν υπάρχει χρήση φυστάμενου δείκτη, όπως είπε και ο Φαμπρίτσιο, αυτό ίως ισχύει μέχρι το 2020, δηλαδή μέχρι την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτος λογικό ε, σαν προσέγγιση, μια διαδοχική προσέγγιση, μια σταδιακή προσέγγιση με την εισαγωγική, με την σταδιακή επιβολή των προϋποθέσεων, των απαιτήσεων και έτσι διευκολύνουμε και τα, την κατάσχετική με τα αιτήματα για άδεια. Γιατί ξέρετε ότι πριν οι δείκτε αναφορά δεν ήταν ρυθμιζόμενοι ε, ρυθμιζόμενο αντικείμενο και άρα χρειάζεται σταδιακά να μπει αυτή η, ιδέα της εποπτείας και ε, του ελέγχου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μια αρχή που δεν έχει ε, ή ένας φορέας μάλλον που δεν έχει αδειοθωτηθεί στο 2020 σημαίνει χωρίς εποπτεία. Πάντα μπορούμε να παρέμβουμε αν υπάρχουν ζήματα παραποίησης στοιχείων δεδομένων εισαγωγής. Για το επόμενο θέμα, πολύ σημαντικό ήταν ε, το καθεστώς των δικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας και οι συνέπειες σε δύο κρίσιμης ε, σημασίας δείκτες αναφοράς με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τη διάχυση των χρηστών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Euribor και αιώνια λοιπόν, πανευρωπαϊκοί δίκτες αναφοράς με συνεισφέρουσες τράπεζες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και χρήστες είτε πρόκειται για χρηματοπιστωτικά μέσα, παράγωγα, υποθήκες, ακόμη και καταναλωτικές συμβάσεις, ε, δια, διάσπαρτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμα σημασίας λοιπόν χαρακτηρίζονται, έτσι πράξαμε, και για το Euribor και προχωρούμε και για το αιώνια. Άπαξ λοιπόν και χαρακτηριστεί ως ε, κρίσιμη σημασία σε ένας δείκτης. Υπάρχει το σύστημα τη συλλογική διαχείριση, υπάρχει το σύστημα της ε, ε, εποπτείας και της υποχρεωτικής συνεισφοράς, που δεν είναι απαραίτητο όμως να χρησιμοποιηθεί, αλλά μένει στο μανίκι σαν ένα ισχυρό μέσο να πιστεί ο συνεισφέρον να συνεχίσει να συνεισφέρει. Και εδώ έρχεται το ερώτημα στη μετατροπή προς το Euribor Plus, όπως εξήγησε νωρίτερα και ο συνάδελφος Φραντσέσκο, η άμεση μετάβαση σε ένα δίκτυο αναφοράς στηριζόμενο στις συναλλαγές δεν ήταν πρόσφορη. Και έτσι ο πάροχος του δίκτυου αυτού αποφάσισε να συνεχίσει με ένα δίκτυο αναφοράς στηριζόμενο σε ε, τιμολόγηση και ορίζοντας ένα υβριδικό, μεικτό δίκτυο αναφοράς. Και εμείς ως νομοθέτης και ως αρχή που προτείνει την νομοθεσία δεν θα παρέμβουμε στο πότε θα γίνει αυτή η μετάβαση, ποια θα είναι η καταλληλότερη στιγμή για τη μετάβαση, θα είναι στα χέρια του ε, παρόχου. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι προσφέρουμε ένα πλαίσιο που συνοδεύει τη μετάβαση αυτή, Euribor τώρα, κρίσιμης αναφοράς δείκτη στο Euribor, θεωρητικά δείκτης αναφοράς ε, που μπορεί να υπαχθεί σε ε, εξουσίες ε, διαχειριστικές όπως και να τον πούμε, αυτό το δίκτυο αναφοράς χαρακτηρίζεται ο Euribor, Euribor Plus κτλ. ως κρίσιμη σημασίας. Και άρα δεν μπορεί να πάψει να είναι Euribor, δηλαδή δεν μπορεί να πάψει να είναι κρίσιμη σημασίας με την αλλαγή του ονόματος σε Euribor Plus. Και άρα τα χαρακτηριστικά παραμένουν και πιστεύουμε ότι οποτεδήποτε και να γίνει αυτή η μετάβαση, όσο χρόνο και αν χρειαστεί αυτή η μετάβαση, ώστε ο διαχειριστής να περάσει από την τιμολόγηση στη συναλλαγή, οπωσδήποτε μένει μέσα στο πλαίσιο το ρυθμιστικό που αφορά τους δείκτες κρίσιμης σημασίας και άρα μπορεί να υπάρχουν οι υποχρεωτικές συνεισφορές ως ε, Συμπληρωματικέ εξουσίες εφόσον δεν υπάρχει ανταπροσωπευτικότητα επαρκής. Άρα σε αυτήν την περίπτωση έχουμε κάνει τη δική μας συνεισφορά για να εξασφαλίσουμε την συνέχεια και πιστεύω ότι αυτό εννοούσατε με την ερώτησή σας τι κάνουμε για να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια των, των δικτών αυτών. Ακριβώς αυτό πω ορίζουμε ότι έχει ο ρυθμιστής, η ρυθμιστική αρχή τα μέσα ανεξαρτήτως του πώς εξελίγεται ένας δείκτης εφόσον είναι κρίσιμη σημασία στηριζόμενο σε τιμολόγηση, σε συναλλαγές θα παραμένει ακριβώς το ίδιο αντικείμενο Euribor που έχει ε, χαρακτηριστεί ως κρίσιμη σημασία. Και ε, το τρίτο, τρίτη μεγάλη ομάδα ερωτήσεων, πάλι πολύ επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικές με την αντιμετώπιση των ε, δικτών τρίτων χωρών, δικτών αναφοράς που παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που έχουν μεγάλη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι μέσω των εκδόσεων χρηματοπιστωτικών μέσων, παραγόγων και χρηματοπιστωτικών συμβάσεων. Εδώ λοιπόν έχουμε τρία μέσα συνέχιση χρήση αυτών των δικτύων αναφορά. Έχουμε το σύστημα τη ισοδυναμία, το σύστημα τη αναγνώριση και το σύστημα τη προσυπογραφή. Για προφανείς λόγους το σύστημα αναγνώρι... ε, ισοδυναμίας όπως λέγαμε, ε, όπως το ονομάζουμε, χρειάζεται μια διαδικασία αναγνώριση από την Επιτροπή. Αναγνώριση ισοδυναμίας. και δεν φαντάζομαι ότι θα ολοκληρωθεί για οποιαδήποτε τρίτη χώρα μέσα στο 2018. Δύο χώρε βρίσκονται σε μια διαδικασία υιοθέτηση κανόνων για του δείκτε αναφορέ, για του διατραπεζικού δείκτε η Ιαπωνία και μάλλον το σκέφτεται και η Αυστραλία. Στο μέλλον θα έχουμε αποφάσεις οδυναμίας που μπορούν βέβαια να υπάρχουν μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση Φερρυπίν ε, στην Ιαπωνία για τους διατραπεζικούς και αντίστοιχα για την Αυστραλία εφόσον προχωρήσει σε αυτήν την ρύθμιση σε ισοδυναμία. Αλλά αυτό, όπως λέω εγώ προσωπικά τουλάχιστον, μπορεί να ε, δούμε να συμβαίνει μόνο στα τέλη του 2018 ή στις αρχές του 2019. Γι' αυτό και ο νομοθέτης, και θα το θυμάστε από τον τριμερή διάλογο, έχει δύο άλλες μεθόδους προβλέψη, που είναι η αναγνώριση και η προσυπογραφή. Και αυτό, υπενθυμίζοντας και τα όσα συνέβησαν ε, στους ε, ε, δείκτες που στηρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε τη δυνατότητα αναγνώριση και προσυπογραφή. Επομένω, με την κατεξουδότηση πράξη κάποιο ο οποίο βγαίνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγει τον κανονισμό ισοδυναμίας και να περάσει μετά, μάλλον τον μηχανισμό ελέγχου για να περάσει μετά επανερχόμενο σε μια αναγνώριση, λόγω τη εγκύτας των δεδομένων αλλά και των λοιπόν κριτηρίων που έχουμε στην καταξουσιοδότηση πράξη, μπορούμε να το εμποδίσουμε εάν υπάρχει μια έκδοση έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη προσέγγισης της εγκύτητας της ε, Πηγέ των δεδομένων ή ε, άλλε ρυθμίσει, τότε περνάμε στο, ε, υπάγεται στο σήμα αναγνώριση ο δείκτης και οι εθνικέ αρχέ θα αναγνωρίσουν το δείκτη αναφοράς ως συνεχιζόμενης χρήσης, μια διαδικασία αρκετά ευέλικτη, πράγμα το οποίο ισχύει λίγο πολύ και για την προσυπογραφή. Δηλαδή, αν πάρει κανείς την άδεια για την προσυπογραφή ενός δείκτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Άρα δεν υπάρχει λόγος άμεσα ανησυχία για το 2019 που να προκύπτει από τους προφανείς λόγους για τους οποίους δεν είμαι σε θέση να ε, εκθέσω περισσότερα επιχειρήματα. Και ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις, ε, ε τις διαπραγματεύσεις είχε αναλάβει η ομάδα Κρούσος, η Task Force. Ε, αλλά τέλο πάντων, όπω και να κλείσουν αυτέ οι διαπραγματεύσει, έχουμε και το σύστημα τη αναγνώρισης, έχουμε και το σύστημα τη προσυπογραφή, που πιστεύουμε ότι θα καλύψουν αυτή την περίοδο μετάβαση και έτσι θα επιτρέψουν στου αρμόδιε αρχέ να αναγνωρίζουν του δείκτε αναφορά για χρήση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να ε, βρίσκουν άλλες αρχές για την προσυπογραφή των δικτών. Βεβαίως μπορεί να περάσουμε μετά περισσότερο σε ένα σύστημα ισοδυναμιών με την προσαρμογή των αντίστοιχων και απαραίτητων αποφάσεων εντωμεταξύ. Αυτά όσον αφορά το ε, σενάριο ε, διάρρηξης, όπως θα το ονομάζαμε, βεβαίως είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην υπάρξει αυτή η διακοπή, η διάρρηξη στην συνέχεια των δικτών. Είμαστε πάντως βέβαιοι ότι ο χρήστης, ο Ευρωπαίος, δεν θα μείνει αποκομμένος από τον, από τον δίκτυο αναφοράς, γιατί αυτό θα είναι εις βάρος όλων μας. Το είδαμε και με τη Euribor και τις συμβάσεις. Αν πάψει να είναι διαθέσιμος ή να υπάρχει ο δίκτυος αναφοράς, αν πάψει να είναι διαθέσιμος γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση, τότε προκύπτει τεράστιο πρόβλημα ως προς την ε, επαναδιαπραγμάτευση ενισχύ συμβάσεων. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να το αποφύγουμε και βεβαίω γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση και οι ανησυχίε που υπάρχουν σε ορισμένε χώρε λόγω μακροχρόνιων συμβάσεων που σχετίζονται με του δείκτε αυτού. Επαγρυπνούμε λοιπόν, έχουμε τα εργαλεία στα θυσία μα. Αν χρειαστεί προσαρμογή του, θα το πράξουμε. Και επίση θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήστη κυρίω δικτών αναφοράς, εξαρτώμεθα από τους δείκτες αναφοράς και από αυτή τη ενία και υπ' αυτή τη ενία υιοθετήσαμε το τρίδημο αυτό των μέτρων, των εργαλείων, για να μην διακοπεί η χρήση και οι συμβατικές σχέσεις, ε, σχέση με τους δείκτες. Και εν τέλει, το ζήτημα των RTS, των ρυθμιστικών τεχνικών προδιαγραφών, Θέλετε μια πρώτη αξιολόγηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι για τις προδιαγραφές αυτές, ε, πώς έχουν ε, λειτουργήσει και αν τις ε, προσυπογράφουμε. Δεν θέλω να κάνω καμιά εκτενή αναφορά στα επιχειρήματα και τις πραγματογνωμοσύνες των ε, ειδικών ε, στα νομικά. Είμαι βέβαιος ότι θα τις προσυπογράψουμε, είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι θα τις προσυπογράψουμε, εφόσον βέβαια τις επαληθεύσουν πρώτα οι νομικές μας υπηρεσίες. Πάντως πρέπει να είναι δυνατόν να γίνει αυτογραφή των RTS. Και εν τέλει θα δημοσιευθούν, για να απαντήσω και στην ερώτηση του Προέδρου, θα δημοσιευθεί το πλήρες κείμενο των ε, δικτών αναφορά. Ελπίζουμε ε, κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας το κείμενο της κατεξουσιοδότησης πράξεως. Διορθώνω. Επομένως το κείμενο θα είναι διαθέσιμο. Αυτό που μπορεί να αναβληθεί και στο συγγνώμη εκ των προτέρων ε, είναι η υιοθέτηση από πλευρά τη Επιτροπή. Θα γίνει δημοσίευση λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτό το παράθυρο των διαβουλεύσεων και θα διατεθεί το κείμενο. Μπορεί όμω η τυπική υιοθέτηση από την Επιτροπή ως Συλλογικό Όργανο, από τους Επιτρόπους δηλαδή, να καθυστερήσει και αυτό το λέω για να διευκρινίσουμε το συγκεκριμένο σημείο. Και επίσης πιστεύω εν τέλει ότι το θέμα που ήγηρε η κόρα και θέλω να μείνω σε ένα σημείο γιατί αναφέρθηκε στις αρχές της ΙΟΣΚΟ της Εθνούς Οργάνωσης. Αυτές είναι ένα σημείο αναφοράς, ένα ορόσημο το ΣΥΠΗΝ για το τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή τι εννοώ ότι μπορούμε, ότι μπορούμε να περάσουμε σε πλήρη ε, υλοποίηση των προδιαγραφών της ΙΟΣΚΟ. Απλώς επειδή υπάρχουν ε, αυτοαποκλεισμοί με τα opt-outs, δεν θα εφαρμόζονται πάντα ομοιό, ομοιόμορφα οι αρχές της ΙΟΣΚΟ. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε και να διορθώσουμε. Επομένω, κοιτούμε τι είδου συνέπειε θα έχουν. Έχουμε τα εργαλεία στη θέσή μα. Και αν δούμε προβλήματα, ασφαλώ σε συνεργασία με την ΕΣΜΑ θα αναστήσουμε και θα υποβάλουμε ευέλικτε λύσεις για το σύστημα της αναγνώρισης από τρίτε χώρε ή τη προσυπογραφή, ώστε να λειτουργήσει το σύστημα πρόσκοπτα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο για να απαντήσουμε. Σε σχέση με το μεταβατικό καθεστώς υπάρχει μια κάποια αβεβαιότητα σε σχέση με τους ισχύοντες ε, κανόνες αναφοράς και τα benchmarks γενικότερα και τους μελλοντικούς. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, άποψή μου, είναι ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει υπόψη το Brexit, αλλά ο κανονισμός νομίζω ότι είναι διαθέσιμο σε αλλαγές μετά από την αποχώρηση της γεκμένης χώρας. Μετά την υιοθέτηση της πρότασης έτσι και αλλιώς το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Και δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα γίνει δεκτό το RTS. Υπάρχει μια κάποια βεβαιότητα χρονική, το ταχύτερο το καλύτερο βέβαια. Η κόρα καταρχάς έχει το λόγο και μετά ίσως ο κ. Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την ΕΣΜΑ και την Επιτροπή που απάντησε στις ερωτήσεις μας. Νομίζω ότι ήταν ικανοποιητικές απαντήσεις στις βασικές μας ανησυχίες θα είναι καλό αν διευκρινιστούν καλύτερα αυτά τα οποία είπατε και αν μας δοθούν γραπτά για τη μεταβατική περίοδο και το πώς ερμηνεύουμε εμείς τα μέτρα αυτά. Καλό θα ήταν να μας το δώσετε γραπτά. Περιμένω λοιπόν να ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα η πρότασή σας για τις κατεξουσιοδότηση πράξης και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία όπως το κάναμε μέχρι τώρα με ένα ανοιχτό και επικοδομητικό τρόπο. Αν υπάρχουν κάποιες περαιτέρω ανησυχίες ή κάποιες σκέψεις ε, και ενούργιες ενημερώστε μας. Θα δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της περίοδου διαβούλευσης. Είμαι επίσης ικανοποιημένη γιατί ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το θέμα είναι ρεαλιστικός εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στρεβλώσουμε τη λειτουργία των αγορών. Εξαρτώμεθα από τα benchmarks και από αυτά μάλιστα που έρχονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε κάνει και την πρόταση για το νέο σύστημα για την επικύρωση και την διαδικασία αναγνώρισης, ακριβώς επειδή υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας αναγνώρισης και αντιστοιχίας. Είναι θέματα αυτά τα οποία ίσως τύχουν περαιτέρω διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Ο κύριος Φερνάντες δεν θέλει το λόγο. Καλώ σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς θα προχωρήσει το RTS. Στόχος για το RTS είναι να το υιοθετήσουμε τρεις μήνες ε, μετά την ε, παραλαβή τους θα τα εξετάσει η νομική υπηρεσία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει γρήγορα. Οι συνάδελφοι νομίζω ότι το είπαν ότι είναι εύκολο να έχουμε τις νομικές απόψεις για τα RTS διότι δεν είναι στην εξουσιοδότηση πράξης. Είναι μια κατηγορία όπου τα πράγματα ελπίζω να πάνε πιο γρήγορα. Okay, but it's uh, next week, so it will be next week. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν δεκτά δηλαδή. Την επόμενη εβδομάδα ε, έτσι και αλλιώς απαιτείται να υπάρξει μια τρίμηνη περίοδος. Θα το κάνουμε αυτό μέσα στο τρίμηνο, λέει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά την αρχική πρόταση για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, τις πέντε κατεξουσιοδότηση πράξεις, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, τρει μήνε δεν είναι μεγάλη περίοδο, λέει ο πρόεδρο. Σα ευχαριστώ όλου για τη συμμετοχή σα. σε μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την υιοθέτηση των κατεξιοδότηση πράξεων. Θα κάνουμε 12 με 15 λεπτά διάλειμμα πριν από τις ψηφοφορίες. Αυτό το οποίο είπατε για τη γραβάτα δεν ισχύει για τα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά θα προσπαθήσω να βρω κι εγώ ένα διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν οι πολιτικές ομάδες και για τα θέματα της παρουσίας.

Dear colleagues, please take seat. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε την ψηφοφορία βέβαια, αλλά και κάποιες ανακοινώσεις πρώτα. Με βάση τον κανονισμό. Δυστυχώς δεν είναι σύντομες ανακοινώσεις, αλλά θα προσπαθήσω να τις πω το δυνατόν πιο γρήγορα. Καταρχάς, ε, σύνομψη αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών ε, με τους διορισμούς. Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ένωση για συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτικών για, Πολιτιών για προληπτικά μέτρα για την ασφάλιση και αντασφάλιση. Προεδρείο και δύο πρόεδρος έλεγχος ε, κεφαλαίων ρευστών που ε, εισέρχονται και αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε σε ποιον θα πάει ακόμα, δεν ξέρουμε σε ποιο άρθρο θα στηριχθεί. Συνεργασία της, ε, των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών, ΙΚΑΡ, σοσιαλιστές γνωμοδότηση, σε αιτήσια έκθεση για τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Προεδρείο για την επαφάση της Επιτροπής Προπολογισμών. Τα υπόλοιπα αναβλήθηκαν. Οικονομική διακυβέρνηση αποφασίζουν οι συντονιστέ να προσκαλέσουν σε οικονομικό διάλογο την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Γαλλία. Θα αποσταλεί σχετική επιστολή στου υπουργού, ανάλογα βέβαια και με, την, ε, με το χρονοδιάγραμμα των υπουργών αυτών θα προσδοριστεί η σχετική συνεδρίαση για να γίνει συνάντηση κατά προτίμηση πριν το καλοκαίρι, κατά πάσα πιθανότητα συζήτηση και στην Ολομέλεια Επίσης αποφασίζουν την αναβολή της αποστολής στη Λισαβόνα για τις 2-3 Νοεμβρίου οι συντονιστέ, εφόσον βέβαια οι συνομιλητές μας είναι ευκαιρία εκείνε τι ημέρε. Επόμενα βήματα για το Brexit. Οι συντονιστέ καλούνται σε πιθανό πρόγραμμα δημόσια ακρόαση ε, εφόσον βρεθεί η κατάλληλη η ημερομηνία. Νοέμβριος, Οκτώβριος-Νοέμβριος. Επίσης ε, θα σταλούν απαντήσεις σχέση με τις αναφορές 0753-088-1217. 19-20 προσοχή συνεδρίαση για, που θα συστήσει τα υπόλοιπα θέματα. Εποπτεία για τον Ιούλιο δεν προβλέπεται. Συντονισμός ε, Βόλου Συμβουλίου θα προσδιοριστεί με την Τζούρι, εφόσον μας το επιτρέπει ο χρόνος, για βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα. Αποφασίζουν οι ομάδες να δώσουν επιπλέον χρόνο για αποστολή στο ΕΛΚ και επιπλέον η Άλντε μπορεί να πάρει μια θέση επιπλέον στην αποστολή στην Πορτογαλία. Ετήματα των πρασίνων μονάδα οίκων αναλαμβάνει την αξιολόγηση των τελευταίων δικτών αναφοράς. Αυτά ως ανακοινώσεις και στις καλές ειδήσει από τον τριμερή διάλογο ολοκληρώθηκαν τρεις τριμερείς διάλογοι με επιτυχία και συγχαρητήρους στους Σύρπα είναι εδώ. Όχι. Πάντως συγχαρητήρια στη Σύρπα Πιετικάινεν για τη θετική κατάληξη του δεύτερου τριμερούς διαλόγου πολύ γρήγορα. Τριμερής διαλόγος για τα κεφαλαία, για τα ταμεία. Πολιτική συμφωνία και ιδιαίτερα σε σχέση με το ρόλο της ΕΣΜΑ. Συμφωνία επετεύχθη. επετεύχθη οι αρμόδιες αρχές θα εξασφαλίσουν ότι η υπαγωγή για την καταχώρηση, η υποβολή των αιτήσεων για την καταχώρηση θα υποβάλλεται στην ΕΣΜΑ και η ΕΣΜΑ θα αναλαμβάνει την επαλήθευση και την εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων, διάθεση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, θα αναπτύξει τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα για την διάθεση των πληροφοριών και γνωστοποίησή τους. Αρχικό κεφάλαιο Euro 50.000, 1.8 ελάχιστες προδιαγραφές κάτω από τις 100.000, περιγραφή περιβαλλοντικών και κλιματικών κινδύνων στην προσέγγιση της ποσοστικοποίησης και της επιχειρηματικής δράσης Μύφιντ επίση για το κεφάλαιο διακινδύνευσης, εισαγωγή και αλλαγή νομικού πλαισίου για την εισαγωγή διαβατηρίου διαχείρισης, εξουσιοδότηση τεχνικό επίπεδο, παραμένει στο κείμενο και η ΕΚΟΝ θα τοποθετηθεί σε προσεχή συνεδρίαση όταν έχει λάβει και τα κείμενα. Ταυτόχρονα Γενική Συμφωνία Πολιτική για τις διασφαλείς συγχαρητήρια στον Οτμαρ Κάρας για την τιτλοποίηση. Πολύ σημαντικό ζήτημα βέβαια για την Ένωση των Κεφαλαιοχικών Αγορών. Συμφωνούμε σε μια καταρχήν ανατροπή της προσέγγισης και βέβαια υπάρχουν παρεκκλήσεις και διαφοροποιημένο καθεστώς για το STS και το non-STS, άρα είναι το όριο. Επιτρέπεται επίπεδο ισότιμης προτιμού ανταγωνισμού και εξασφαλίστη τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Διαφυλάσσεται η τιτλοποίηση, με με τζανίνα διαφυλάσσονται οι κανόνες για το επίπεδο 5% έναντι της εισαγωγής της προϋπόθεσης αποκάλυψης των κινδύνων και υποχρέωση για την Επιτροπή της Γνωστοποίησης ή ονδήποτε κινδύνων μπορεί να προκύψουν σε εγκάρσια ή οριζόντια επίπεδα, επαλήθευση για τους εκδότες εάν τηρούν τις προϋποθέσεις τιτλοποίησης και σημαντικές προϋποθέσεις ελέγχου για τον εκδότη. Ο συνεισηγητής διατηρεί το EPA για τις κατευθυντήριες γραμμές, την ε, EBA, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, για τα κριτήρια, καθυστέρηση επίσης μέχρι τις 18 Ιουλίου κάποιων μηνών ώστε να υπάρξει δυνατότητα προσαρμογής για τους μάρκες, για τους ε, συμμετέχοντες στην αγορά και ένα και για την ανάπτυξη ενός πιο στεναρού μακροπροληπτικού πλαισίου. Με σημαντικές επιτυχίες πάντα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα αυτά τεχνική δουλειά που έχει ολοκληρωθεί και οδηγεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στην έγκριση του ελληνικού κειμένου με βάση ιστορικές διαδικασίες στις προσεχείς εβδομάδες. Και εν τέλει ολοκληρώσαμε, αλλά θα είμαι πιο σύντομος εδώ, το τριμερή διάλογο για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα. Σχέδιο κανονισμού. Διάφορες πτυχές, στατιστική κάλυψη της φτώχειας, μεταναστευτικές ροές, χάσμα φύλου, επικαιρότητα κατάθεσης και ποιότητα δεδομένων, θέσεις δηλαδή του Κοινοβουλίου, δύο τριμερείς διάλογοι. Για το ΕΦΣΙ μετά από δύο τριμερείς διαλόγους ε, είχαμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε όλες τις θέσεις αναλυτικά για, περισσότερα τα για τα περισσότερα από τα πολιτικά θέματα και στο δεύτερο τριμερή διάλογο έγινε προπαρασκευαστική εργασία από την Κομισιόν που επέτρεψε παραγωγική συζήτηση για θέματα που έχουν να κάνουν προστατικότητα, την τιμολόγηση, το δίκτυο αποτελεσμάτων, τον πίνακα αποτελεσμάτων και την φορολόγηση. Έχουμε καταλήξει σχεδόν σε ορισμένα θέματα, αλλά ορισμένα άλλα πρέπει ακόμη να συζητηθούν όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση. Ο επόμενο τριμερή διάλογο θα γίνει στις 12 Ιουνίου το βράδυ στο Στρασβούργο. Ο τριμερής διάλογος για τα μέτρα κατά της ε, νομιμοποίησης ε, του προϊόντος εγκλήματος ε, συζητήσαμε τα θέματα πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους και ζητήσαμε από το Συμβούλιο να υπάρχουν οι αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις για να υπάρχει πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία δικαιούχων των εταιριών, τους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πρώην πολιτικούς και γενικά το καθεστώς ε, καταπολέμησης της κατάστασης αυτής και ιδιαίτερα για το Μητρό των ε, χωρών ε, υψηλού κινδύνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται.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 Thank you. Okay. Οπότε. Μετά τη σοφορία. Α, πριν. Παρακαλώ. Μία πολύ σύντομη δήλωση της εισηγήτριας, η κόρα. Ευχαριστώ από πλευράς του συγητή κυρίου Τόιερ που δεν μπορεί να παρευρεθεί δυστυχώς. Ο συγητής ευχαριστεί τους συναδέλφους για την επικοδομητική συνεργασία για την πρόοδο που επιτεύχθηκε. Θεωρεί ότι οι συμβαστικές ε, είναι μια αντικειμενική απεικόνηση του τρόπου σκέψης των συναδέλφων. Υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ των ε, σκιωδών ότι οι προθεσμίες θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόδοξες. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Οι εθνικές αρχές συχνά δεν έχουν επαρκή κίνητρα για να δράσουν σύντομα και να επιλύσουν τις διαφορές διπλής φορολόγησης, όπως αποδείχθηκε από υποθέσεις που διαρκούν πάνω από δύο χρόνια. Άρα υπάρχει σοβαρή δυνατότητα και περιθώριο βελτίωσης. Γι' αυτό προτείνουμε να επιταχυνθούν οι διάφορες φάσεις διαδικασίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αφιερώνουν επαρκές ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Χρειάζεται αποτελεσματικό σύστημα φορολόγηση των εταιριών που θα επιτρέψει τι εταιρείε να αποφελθούν πλήρω από την ενιαία ώρα. Ευχαριστεί όλου που συμμετείχαν για τη στήριξη και τη συμβολή του. Και φυσικά μεταξύ αυτών είναι η γραμματεία τη ΕΚΟΝ και οι Σκιώδη. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Να ψηφίσουμε τώρα. Τροπολογία 85 υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Σεβαστική Α. Υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 149 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται. Αν θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 173 και 4 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται εγκρίνεται με μία ψήφο πλειοψηφία 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά και εδώ να ελέγξουμε. Βλέπω μερικούς πολύ ενδιαφέροντες και πρωτότυπους συνδυασμούς πολιτικών ομάδων και μεταβαλλόμενους. S&D, ECR, Πέρας. Απορρίπτεται. 178. Ε, συγγνώμη, συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ΚΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά εγκρίνεται 31 γιατί η προηγούμενη καταπίπτει υπέρ κατά εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, απορρίπτεται συγγνώμη 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, πηδήξαμε την 178. Με συγχωρείτε. Στη σελίδα 12 του καταλόγου Σοφοριών λοιπόν. 178 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Την 178 άρχεται. Δύο συνάδελφοι δεν ψήφισαν ακόμη. Πέρας. Πέρας λέγω. Απορρίπτεται. Λοιπόν, 33 αν θυμάμαι καλά για τις ιδεολογικέ αναφορέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά απο... Α, να ελέγξουμε. Τη 42. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο επιπλέον. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 79 άρχεται πέρας απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 81 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Η, η 7 και 82 καταπίπτουν. 83 λοιπόν υπέρ κατά Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα την τροποποιηθήσα πρόταση της Επιτροπής. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 41 ψήφους και μία ψήφο κατά και μία αποχή. Α, υπάρχει μία τροπολογία για το νομοθετικό ψήφισμα καινοτόμως διαδικασία. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας την ελέγξουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Λοιπόν, το νομοθετικό ψήφισμα ενεκρίθη όπως τροποποιήθηκε. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε γιατί έχουν αλλάξει οι κανόνες στον εσωτερικό μας κανονισμό να συγχαρούμε τον εισηγητή. Okay, so uh, next uh, meeting, but before that, allow me uh, Κάτι το προσωπικό. Θέλω να ευχαριστήσω και να ευχηθώ ότι καλύτερο στη Λάουρα Φορμιζάνο, η οποία εγκαταλείπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια όλο αυτό τον καιρό.